είτε και εμείς είμαστε στο πλευρό του και εκφράζουμε την ελεγγύη του. Έρχομαι στι ανακοινώσει. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στις 10 Φεβρουαρίου έγκρισε ε, ενέκρινε συγγνώμη, ε, την εντολή της κυρίας Ρίνα Ρόνια Κάρη και πρότεινε να εγκριθεί ε, από 5η Φεβρουαρίου 2014. Προτείνω να ε, θεωρήσουμε έγκυρη την εντολή αυτή. Έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις, όχι. Οπότε διαπιστώνεται η εγκυρότητα της εντολής της κυρίας Κάρη. Οι αρμόδιες επιτροπές έχουν κάνει διορθώσεις